Okay, friends. Ε, Αγαπητοί φίλοι, προχωράμε στη συνεδρίασή μας. και χαίρομαι που έχουμε του εκπροσώπου τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρώτο όμως ένα μήνυμα από του Διερμηνεί. Βρισκόμαστε ήδη στην 38η μέρα των ε, κινητοποιήσεων λόγω τη άδική επιβολή ε, από τη δίκη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εργασιακών, ε, της μονομέρους επιβαλής άδικων εργασιακών συνθήκων. Γι' αυτό το λόγο η, η διερμηνία θα διακοπεί στις 12.30 ακριβώς, δηλαδή την προβλεπόμενη ώρα λήξης της συνεδρίας. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση. Θα ακούσουμε λοιπόν την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα μας παρουσιάσει την πρόταση για το ενισχυμένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Είναι σημαντικό αυτό το θέμα για μας, γιατί πολλά ζητήματα αρμοδιοτήτων μας ε, αφορούν το ταμείο αυτό. Και ο κανονισμός που πραγματεύεται θέματα που μας ενδιαφέρουν είναι πολύ σημαντικός για την Επιτροπή μας. Γιατί μην ξεχνάτε ότι είμαστε Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Δίνω το λόγο λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας κάνει την εισαγωγή. Ευχαριστώ και στην Προεδρία μάλλον. Ευχαριστώ. Καταρχήν να σας δώσω μερικά γενικά σχόλια του ιστορικού και ποιες προκλήσεις προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε την πρόταση. Καταρχήν, ζούμε σε έναν κόσμο που η τεχνολογία η παραγωγικότητα και η παγκοσμιοποίηση επηρεάζουν κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας. Θα πρέπει λοιπόν να αναβαθμίσουμε τις δεξιότητες του εργατικού δυναμικού για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, των τεχνολογικών εξελίξεων και της ψηφιοποίησης, αλλά και να δημιουργήσουμε μια οικονομία υψηλής ανθεκτικότητας και χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Η κατάσταση της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βελτιωθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια, αλλά εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε σημαντικές, σημαντικά ποσοστά μακροπρόθεσμης ενέργεια και κυρίως ενέργεια των νέων. Αυτές οι τάσεις είναι πολύ ανησυχητικέ και εξακολουθούν να ισχύουν σε αρκετά κράτη-μέλη. Υπάρχουν βέβαια μεγάλες διαφορές και ανισότητες επίσης μεταξύ των κρατών μελών. Εξού και η ανάγκη να αντιμετωπίσουμε κυρίως το ζήτημα της ενέργεια των νέων που παρά την μείωση του από τον Ιανουάριο του 2013 που είχαμε 24% κοινοτικό μεσόωρο ανθρώπων που δεν είχαν απασχόληση ή δεν παρακολουθούσαν καμία σπουδή κατάρτιση και το 2018 είναι 15,6% το Μάρτιο του 2018, έχουμε αισθητή μείωση 5% περίπου, αλλά σε κάποιες χώρες μέλη έχουμε και πολύ ψηλότερο ποσοστό ανεργία των νέων ή που δεν παρακολουθούν σπουδέ ή οποιαδήποτε άλλη μορφή κατάρτιση. Αλλά αν συγκρίνουμε το ποστό ενεργείας των νέων σε σχέση με το γενικό συντελεστή ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπουμε ότι το ποστό ανεργίας των νέων είναι διπλάσιο από την ανεργία του υπόλοιπου εργατικού δυναμικού. Θα πρέπει λοιπόν να σπυρώσουμε τις δυνάμεις μας και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μειώσουμε τον αριθμό των νέων που δεν έχουν θέση εργασία ή δεν παρακολουθούν σπουδέ ή οποιαδήποτε κατάρτιση και να εξασφαλίσουμε ένα πιο ευήμερο μέλλον για όλου. Δεύτερη πρόκληση αφορά την κοινωνική κατάσταση στην Ευρώπη. Ε, πολλοί ε, βρίσκονται σε, ε, στα καταφύλλα τη φτώχεια, Βέβαια, μεταξύ 2012 και 2015 είχαμε μείωση κατά 4,8 εκατομμύρια των ανθρώπων αυτών. αλλά το 2016 118 εκατομμύρια συνάνθρωποι μας βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχεια ή κοινωνικού αποκλεισμού, κάτι που δείχνει πόσο μεγάλες κοινωνικές ανισότητες υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών. Επίσης, ε, ακόμη και στο εσωτερικό των χωρών υπάρχουν ε, μεγάλες διαφορές. Η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός ε, αυξάνεται στα αστικά κέντρα των 15 χωρών και στις 13 νέες χώρες μέλη και την Κροατία που μπήκαν μετά το 2004, ο αγροτικός πληθυσμός αντιμετωπίζει μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού από τον αστικό πληθυσμό. Μια άλλη πτυχή αυτών των κοινωνικών ανισοτήτων και της περίπλοκης κοινωνικής κατάστασης είναι ότι μερικές ε, ομάδες μειονοτήτων επηρεάζονται δυσανάλογα από τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και ένδυας. Και αυτή την πρόκληση λοιπόν θα πρέπει να την αντιμετωπίσει το ενισχυμένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Και επίσης έχουμε μια άλλη πρόκληση πολιτικής που αφορά τις δημογραφικές ε, τάσεις ο πληθυσμός γυράσκει, οι εργαζόμενοι είναι όλο και πιο ηλικιωμένοι και επίσης έχουμε αυξαμένο ρυθμό υπηκών τρίτων χωρών που έχουν λάβει άδεια διαμονής και εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεταξύ του 2014 και του 2017 μάλιστα είχαμε 1,7 εκατομμύρια υπηκών τρίτων χωρών που έλαβαν άδεια Διαμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να αναπτύξουμε πολιτικές ένταξης στην αγορά εργασίας για όλους αυτούς τους υπηκόου τρίτων χωρών ε, που ήδη είναι μετανάστες ή ή είναι μέλη μειονοτικών κοινοτήτων για να έχουμε ευκαιρία στην αγορά εργασίας. Έτσι θα καταπολεμήσουμε τις ανισότητε, τις διακρίσει και θα εξασφαλίσουμε ίσε ευκαιρίε για όλου. Σε ό,τι αφορά το, την πολιτική, το πολιτικό υπόβαθρο της πρότασης, έχουμε την 60η επέτειο της ε, ίδρυσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και πέρυσι το Μάρτιο στη Ρώμη οι ηγέτες 27 χωρών μελών και κοινοτικών θεσμικών οργάνων υπέγραψαν το θεματολόγιο της Ρώμης και υποσχέθηκαν ε, να εντείνουν τις προσπάθειές τους για μια πιο κοινωνική Ευρώπη. Και αυτό είναι ο φάρος για τις πολιτικέ μα. και μάλιστα έχουμε εκδώσει μια λευκή βίβλο για το μέλλον τη Ευρώπη με πέντε έγγραφα πολιτική, έγγραφα προβληματισμού για να τροφοδοτήσουμε τη συζήτηση για το πώ θέλουμε να αναπτυχθεί το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τον Νοέμβριο ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων ε, υπευλήθη στην Σύνοδο Κορυφής του Γκέτεμπορκ και αυτός ο πυλώνας, Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων ε, έχει πια περιληφθεί στο δημόσιο λόγο όλων των κοινοτικών θεσμικών οργάνων που ε, ασχολούνται με θέματα απασχόλησης ε, και πάταξης του κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτό είναι πραγματικά μία από τις πηξίδες των πολιτικών μας προκειμένου να έχουμε πιο δίκαιες και ίσες ευκαιρίες για σπουδές, κατάρτιση και απασχόληση. Και οι αρχές και τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων συνάδουν με τους ε, στόχους βιώσιμης ανάπτυξης ε, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από το 2015. Στις 2 Μαΐου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε το νέο πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027. Και με την πρότασή μας αυτή για το επόμενο ΠΔΠ ε, εντοπίζουμε ξεκάθαρα τους πόρους που προτείνουμε και τα κονδύλια για το ενισχυμένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Ε, περίπου 112 δις με τρέχουσες τιμές. Έχουμε όμως και ένα άλλο ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, το οποίο γνωρίζετε ιδιαίτερα στην Επιτροπή σας, που ε, βρίσκεται εκτός του μελλοντικού πι και θα έχει αυξανόμενο ανώτατο όριο ετήσια ικανότητα για να κινητοποιήσει κονδύλια ύψου 225 εκατομμυρίων το χρόνο. 150 είναι, εκατομμύρια το χρόνο είναι το ισχύον ανώτατο όριο. Αυτά με λίγα λόγια είναι η δομή του προϋπολογισμού του ΕΚΤ Plus, του ενισχυμένου ή διευρυμένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Επίσης, τα ε, και δις ε, του ενισχυμένου ΕΚΤ που θα επενδύουν άμεσα στο, στο ανθρώπινο δυναμικό στην επόμενη πηδελταπή δίνει μια πιο φιλόδοξη διάσταση στο μελλοντικό πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Το ενισχυμένο ΕΚΤ ε, θα ακολουθήσει τρεις τρόπους διαχείρισης. Καταρχήν την επιμερισμένη διαχείριση. Εκεί τα κράτη-μέλη θα συνεχίζουν να ετοιμάζουν τα προγράμματά τους και να δίνουν τα κονδύλια με βάση τι προτεραιότητες Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και τις ε, προτεραιότητες που περιλαμβάνονται στις στάσεις αναχώρα και στις ε, ε, επενδυτικούς προανατολισμούς του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ε, βέβαια, έχουμε μειωμένα, μειωμένες απαιτήσεις συγκέντρωσης τώρα για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις μας θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα της κοινωνικής ένταξη, της καταπολέμησης, της εξάλληψη τη φτώχεια, και γι' αυτό προτείνουμε 25% τουλάχιστον του ενισχυμένου ΕΚΤ ε, στα πλαίσια της επιμερισμένης διαχείρισης να αφιερωθεί σε μέτρα που θα στηρίξουν την κοινωνική ένταξη των χρηζών βοηθείας. Και τουλάχιστον 2% της σχετικής υποστήριξης θα πρέπει να πηγαίνει άμεσα στους απόρους συνεχίζοντας τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Παροχής Βοήθειας στους Απόρους στα πλαίσια της τρέχουσας δημοσιονομικής περίοδου. Η κατάσταση των νέων που δεν έχουν εργασία, δεν παρακολουθούν σπουδέ ή κάποια κατάρτιση, έχει ειδικά κονδύλια Οπότε και το θέμα της συγκέντρωσης ε, αφορά τα κράτη-μέλη, όπου το επίπεδο των αναγκών ξεπερνάει τον κοινοτικό μεσόρο και αυτά τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αφιερώσουν τουλάχιστον 10% του ΕΚΤ ε, στα πλαίσια της επιμερισμένης διαχείρισης για μέτρα που θα βοηθούν τους νέους <clears throat> που δεν παρακολουθούν σπουδές κατάρτιση ή δεν έχουν θέσει εργασίας για να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, να έχουν κάποιες ευκαιρίες να βρουν δουλειά ή να ξεκινήσουν τις δικές τους επιχει... επιχειρήσεις. Βέβαια, αυτό το 10% δεν αποκλεί τα υπόλοιπα κράτη-μέλη που δεν έχουν τόσο υψηλό ποσοστό ενεργείας νέων πάνω από το κοινοτικό μέσο αλλά μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια αυτά για να στηρίξουν τους νέους με ειδικά μέτρα. Για πρώτη φορά το ενισχυμένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προβλέπει ειδικά κονδύλια για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τις αεροκατοικημένε περιοχές. 400 εκατομμύρια είναι η πρόταση. Ε, μάλιστα πέρυσι στην ανακοίνωσή μας ε, είχαμε αναγνωρίσει τις εξόχως απόκεντρε περιοχέ ω ιδιαίτερα ε, μειονεκτούς περιοχές λόγω της απόστασης και είπαμε ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν μέτρα αντίστοιχα με αυτά που ισχύουν για τις χώρες της περιφέρειας της Ευρώπης. Επίσης, το θέμα της ε, διεθνικότητας, ε, διακρατικότητας, 200 εκατομμύρια, είναι τμήμα ε, της εφαρμογής στα πλαίσια της επιμερισμένης διαχείρισης. Οι δραστηριότητες αυτές διακρατικότητας τη χάνουν κεντρικής διαχείρισης. προτείνουμε 200 εκατομμύρια κονδύλιο για τέτοιου είδους δραστηριότητες που θα συνδέονται με την άμεση διαχείριση για την απασχόληση και την κοινωνική ε, καινοτομία. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε ετήσια προγράμματα, αλλά και πολυετή, με συγκεκριμένους όμως στόχους και πολύ συγκεκριμένη στοχοθέτηση. Ήδη ξεκίνησα ε, με έναν άξονα άμεσης διαχείρισης που είναι το θέμα της απασχόλησης και της κοινωνικής καινοτομίας και για να έχουμε καλύτερη συνέργεια και συμπληρωματικότητα αλλά και συνοχή όλες οι άμεσες ενισχύσεις στο εργατικό δυναμικό και στο ανθρώπινο δυναμικό ε, θα καλύπτουν και το θέμα της ε, υγείας που θα υπόκειται στην άμεση διαχείριση με ισχυρή ανάμειξη των συναδέλφων της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και με τη συνεχή εφαρμογή συγκεκριμένων στόχων και ομάδων στόχων που εντοπίσαμε στην τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού. Αυτή είναι μια επισκόπηση των πέντε ταμείων που θα συνενωθούν στα πλαίσια του ενισχυμένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Μάλιστα, προσεγγίζουμε τη νέα περίοδο προγραμματισμού με κάποιους πρωταρχικού στόχους. Καταρχήν θέλουμε να εξασφαλίσουμε τη συνοχή και τη συνέργεια μεταξύ των ταμείων που συμβάλλουν άμεσα στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Επίσης θέλουμε να πλουστεύσουμε τη δομή του και να διευκολύνουμε τους χρήστες και δικαιούχου των ταμείων να εντοπίσουν ε, τις ε, χρηματοδοτικές ε, δυνατότητες που έχουν στα πλαίσια της τρέχουσας περίοδου ε, σε σχέση με τις προκλήσεις και κάνουμε σχετικές μελέτες επιπτώσεων και άλλες εκθέσεις και προσπαθούμε να διευκολύνουμε όσο μπορούμε τους δικαιούχους να εντοπίσουν σε ποιου τομεί μπορούν τα προγράμματά τους ε, οι ιδέες τους ε, να τύχουν υποστήριξης. Επίσης θέλουμε να μειώσουμε τον αριθμό των προγραμμάτων και νομίζω ότι με την συγχώνευση πέντε ταμείων καταφέραμε να συνεισφέρουμε στην γενική μείωση των προγραμμάτων στο τωρινό και στο μελλοντικό ΠΔΠ. Τώρα έχουμε 48, στο μέλλον θα έχουμε 37 τέτοια προγράμματα, οπότε υπάρχουν πολλές συνέργειες και πολλή προσπάθεια που μπορεί να γίνει και να βελτιωθεί ε, αν είναι όλα εντός του ιδίου νομικού πλαισίου. Και τέλος όλα αυτά θα συνεισφέρουν στο να υλοποιούν τις αρχές του κοινωνικού πελώνα στα κράτη-μέλη. Όλα αυτά θα συνεισφέρουν σε 11 συγκεκριμένους ε, στόχους που σχετίζονται με τις αρχές και τα δικαιώματα του πυλώνα. Εδώ και πάλι έχουμε μια γενική παρουσίαση για να δούμε ακριβώς που βρίσκονται τα ταμεία με την κοινή διαχείριση, την άμεση διαχείριση στον κανονισμό Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ. Θα ήθελα τώρα να ξεκινήσω. Έχουμε κάποιες αναθεωρήσεις ε, που βρισκόταν πριν σε τέσσερις κανονισμούς. Προσπαθήσαμε λοιπόν να δούμε τους συγκεκριμένους στόχους, αρχές και ιδιαιτερότητες του Ευρωπαϊκού Ταμείου να μπουν όλα σε έναν κανονισμό. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι οι κανόνες εφαρμογής γενικά βρίσκονται στον κανονισμό των κοινών διατάξεων. Ο κανονισμός ESFC ε, έχει κάποιες ιδιαιτερότητες για τις επενδύσεις στους ανθρώπους και στους συγκεκριμένους στόχους που θα πρέπει να ισχύουν για όλες τις δέσμες ε, του κανονισμού και για όλες τις δραστηριότητες ε, που στηρίζει το Ταμείο. Η γενική στόχη λοιπόν όλων των δεσμών αυτών είναι να στηρίξουμε την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, ενώ οι δέσμοι της κοινή διαχείριση λαμβάνουν υπόψη και τις κατευθύνες γραμμές απασχόλησης και τις συστάσεις αναχώρα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Η δέσμη κοινωνικής καινοτομία και απασχόλησης εστιάζει στην κοινωνική προστασία, ένταξη, εργασιακέ συνθήκες, απασχόληση και το κομμάτι της υγείας θα συνεχίσει την κατεύθυνσή του για να διασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συγκεκριμένοι, 11 συγκεκριμένοι στόχοι του κανονισμού υπάγονται σε έναν στόχο του κοινού κανονισμού για να δημιουργηθεί μια πιο κοινωνική Ευρώπη και προβλέπει δραστηριότητες ε, στον τομέα της απασχόλησης, εκπαίδευσης, ε, κοινωνικής ένταξης και της υγείας. Γίνονται συγκεκριμένες αναφορές ε, στους μετανάστες και σε κάποια βασική ηλική βοήθεια που εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή και πρέπει να ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο του κανονισμού Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ και θα πρέπει επίσης ε, να συνεισφέρει και σε στόχους ε, άλλων κατευθυντήριων γραμμών του κανονισμού για μια έξυπνη Ευρώπη και μια πράσινη Ευρώπη για να γίνει η οικονομία μας πιο πράσινη. Οι συγκεκριμένοι στόχοι μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις ομάδες. Έχουμε τους τρεις συγκεκριμένους στόχους που αφορούν τον στόχο της απασχόλησης. Θέλουμε δηλαδή να έχουμε ευκολότερη πρόσβαση στην δουλειά για όλους, να εξυγχρονιστεί η λειτουργία της αγοράς εργασίας και θέλουμε συγκεκριμένα να στηρίξουμε τη συμμετοχή των γυναικών, να υπάρχει ισορροπία με την οικογενειακή ζωή, να υπάρχουν ε, οι δυνατότητες για τη φροντίδα των παιδιών, για να μπορούν οι γυναίκες να πάνε στη δουλειά και να έχουμε κάποιες δραστηριότητε οι οποίες θα προσαρμόζουν το χώρο εργασίας ε, στους ε, εργαζόμενους, στους ηλικιωμένους εργαζόμενους, στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης τώρα. Επίσης υπάρχει ανάγκη για καλύτερη ποιότητα των συστημάτων εκπαίδευση και κατάρτισης, την ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση και κατάρτιση σε όλους και την ανάγκη επίσης επανεκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης των ανθρώπων λαμβάνοντας υπόψη τις ψηφιακέ δεξιότητε που θα απαιτούνται στο άμεσο μέλλον. Επίσης έχουμε συγκεκριμένο στόχο για τις αλλαγές σε επίπεδο εταιρείε, αλλά και τις απαιτήσει ε, ε, που πλέον αφορούν και άτομα τα οποία ήδη έχουν κάποια δουλειά. Στον τομέα της κοινωνικής ένταξης θέλουμε με ενεργά μέτρα ένταξης θέλουμε να έχουμε την δυνατότητα να εντάξουμε τους μετανάστες υπηκόους τρίτων χωρών και κοινότητες όπως η Ρωμά θέλουμε να συνεχίσουμε να παρέχουμε πρόσβαση σε ποιοτικέ ε, βιώσιμες υπηρεσίες, συστήματα κοινωνικής προστασίας, ε, αποτελεσματικότητα και αντοχή των συστημάτων υγείας και μακροπρόθεσμης ε, φροντίδας και επίσης ένταξη των πιο αποκλεισμένων. Θα ήθελα να τονίσω τις οριζόντιες αρχές που σχετίζονται με την ε, ένταξη στοχευμένων δράσεων για να υποστηρίξουμε την ε, ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τις ίσες ευκαιρίες και να αποφύγουμε τη διακριτική μεταχείριση. Θα συνεχιστεί η δυνατότητα για να υπάρξει αποϊδρυματοποίηση και να περάσουμε σε μια φροντίδα στι οικογένειε και εντός της ε, κοινότητα και πρέπει να συνεχιστεί αυτό, έχει ξεκινήσει εδώ και κάποια χρόνια. Πολλέ ε, πολιτικές ε, και προσοχή αποδίδεται σε αυτό έτσι ώστε άτομα με προβλήματα, με αναπηρία να αισθάνονται μέλη της κοινωνίας. Γίνεται τι επίσης αναφορά στο ότι δεν θα στηρίζουμε κάποια δράση που θα συνεισφέρει στον κοινωνικό αποκλεισμό και τον διαχωρισμό. Αυτά θα είναι στοιχεία όλης της διαδικασίας ε, επιλογής ε, όταν επιλέγουμε έργα. Έχουμε κοινέ διατάξει ε, για τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού ε, Κοινωνικού Ταμείου ε, ΣΥΝ. Να εφηγαμιστεί περισσότερο με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και τον πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Έχουμε προβλέψει μεγαλύτερη ευελιξία και θεματική συγκέντρωση. Τα κράτη-μέλη θα θέσουν το πολύ, ε, είχαν πέντε επενδυτικές προτεραιότητες, τώρα έχουμε δύο απαιτήσει ε, προσημείωσης για υποστήριξη στα κράτη-μέλη. Με μεγάλη ενεργεία των νέων ή με κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Η με κινδυνο φτωχειας και κοινωνικό χρηματοδότηση είναι κάτι που θα αποφασιστεί από τα κράτη-μέλη σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διαπραγματεύσεις και σε σχέση με τις συστάσεις αναχώρα αλλά και σε σχέση με τα διάφορα προβλήματα και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Ε, στον ε, κανονισμό αυτό εξετάζουμε τη δυνατότητα ε, να ε, δούμε τι γίνεται με τη βοήθεια στους απόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδική προτεραιότητα με πιο απλούς κανόνες εφαρμογής και υλοποίησης. Τα προγράμματα που τρέχουν ε, σήμερα θα συνεχιστούν. Επίσης, χρειάζεται υλικοτεχνικός εξοπλισμός, οχήματα κλπ. Ε, και έχουμε προσπαθήσει να μειώσουμε τους δείκτες, να απλουστεύσουμε τις διαδικασίες. Οι δείκτες ενδεικτικά από 44 έχουν μειωθεί σε 23 και τα κράτη-μέλη ε, καλούνται να χρησιμοποιήσουν διοικητικά μητρώα ε, όταν κάνουν τις κοινοποιήσεις και τις αναφορές τους και με κοινού δείκτες να αναφέρουν στοιχεία για τους δικαιούχους. Με αυτές τις απλοποίησεις ελπίζουμε η εφαρμογή, ε, η εκτέλεση και ο έλεγχος του προγράμματος να είναι πιο εύκολος. Η θεματική συγκέντρωση τώρα ε, είναι ε, ότι ψάχνουμε κάθε φορά το κατάλληλο ποσό για να υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη και τα προβλήματα που έχουν στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και στις συστάσεις αναχώρα ε, υπάρχουν επενδυτικές ε, κατευθύνες γραμμές. Επίσης, ε, προβλέπουμε ευθυγράμμιση για την αρχή και το μέσο της περίοδου με βάση το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για το 2019 και το 2024. Θα υπάρξει μια ενδιάμεση ε, αξιολόγηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου, των προτεραιοτήτων, των προβλημάτων και των αναγκών των κρατών μελών για να ανταποκρινόμαστε καλύτερα σε μεταβαλλόμενες ανάγκες. Υπάρχουν και άξονες προτεραιότητας ε, και είναι πιο εύκολο έτσι να ελέγχεται ε, η υλοποίηση. Μίλησα πολύ για τη θεματική συγκέντρωση. 25% ε, αφιερώνεται ε, στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και στην κοινωνική ένταξη και το τουλάχιστον 2% για τους πλέον απόρους για να συνεχιστεί το πρόγραμμα στο μέλλον. Στο έκτες είναι έχουμε προβλέψει και πιο ομαλή μετάβαση των πλέον απόρων και μειονεκτούντων, εκείνων που έχουν σοβαρέ ε, υλικέ ε, ανάγκες και προβλήματα, για να βγουν από αυτή την κατάσταση και να έχουν ε, πρόσβαση στην εργασία, στην κατάρτιση, στη μετακπαίδευση και μέσω του ΕΚΤΣΙΝ αλλά και άλλων μέτρων για την κοινωνική ένταξη που ήδη έχουμε εντοπίσει και ταυτοποιήσει στα προγράμματα των κρατών μελών. Τρίτο στοιχείο της θεματικής συγκέντρωσης, να δίνεται 10% στους νέους, ε, τους needs, που είναι εκτός εκπαίδευσης, ε, κατάρτισης εργασίας. 15% προτείνουμε για τις πιο απομακρυσμένες περιοχές, στη περιφερική χρηματοδότηση, ακριβώς για αυτούς τους νέους. Είναι αυξημένο το ποσοστό γιατί είναι και μεγαλύτερες οι προκλήσεις λόγω ε, της απόστασης από την εδώ χώρα, από την υπηρετική χώρα. Και ε, λόγω μεταφορικού ισοδύναμου. Είναι σημαντικό να έχουμε ένα ειδικό κονδύλι για τους νέους needs για να ε, συνεχιστεί η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων και στο ΕΚΤΣΙΝ για να αποφευχθούν κάποια προβλήματα που είχαμε ε, εντοπίσει στην τρέχουσα περίοδο. Είναι πιο δύσκολη η παρακολούθηση, ε, ο προγραμματισμός κτλ. Γιατί είχαν ξεχωριστό προϋπολογισμό που έπρεπε να συνδυάζεται με τα κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Και αυξάνοντα το κονδύλι για τους ε, νέους νίτς, ε, καλούμε τα κράτη-μέλη να επαναπρογραμματίσουν πολλά ΕΣΠΑ, έτσι ώστε να υπάρχει σωστή χρηματοδότηση. Αυτά άλλωστε έχει συστήσει και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Ότι είναι τεχνητό ο διαχωρισμός του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και της πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων. Είναι από τα βασικά στοιχεία για την εγγύηση για την νεολαία αυτό. Μέχρι τώρα αυτό το μέσο υποστηρίζει με μονομένες ατομικές περιπτώσεις, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μπορεί να χρηματοδοτήσει ε, διαρθρωτικές αλλαγές, ε, εξατομικευμένες υπηρεσίες στα κράτη-μέλη. With Uh, και ελπίζουμε με τον προγραμματισμό ε, αυτών των ε, πιστώσεων κατά προτεραιότητα θα μπορούμε καλύτερα και να ελέγχουμε και να αναφέρουμε τα επιτεύγματα και τα αποτελέσματα αυτών των μέτρων. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ και τα άλλα ευρωπαϊκά ταμεία. Εδώ υπάρχει ένα άρθρο 7.1, είναι πολύ σημαντική η σχέση Υπάρχουν κάποια προαπαιτούμενα που ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να εξασφαλίσουν το συντονισμό, τη συμπληρωματικότητα και τη συνοχή των ε, διαφόρων ταμείων για να μην υπάρχουν επικαλύψεις ή δυνατόν. Και σε επίπεδο κρατών μελών υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη ακριβώς να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των αρχών που διαχειρίζονται διάφορα ταμεία. Παράδειγμα, άσυλο, ε, μετανάστευση και ένταξη, το ταμείο αυτό το ΑΜΙΦ στα κράτη-μέλη και τα προγράμματα του Κοινωνικού Ταμείου δεν συνεργάζονται πάρα πολύ στενά. Ε, πρέπει ε, οπωσδήποτε να ε, δρομολογούνται από κοινού αυτές οι δραστηριότητες από την αρχή, από το προγραμματισμό, έτσι ώστε είναι που αυτή τη στιγμή υποφελούνται από το ΑΜΙΦ να περάσουν απρόσκοπτα στη χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ. Επίσης, Θέλουμε σε όλα τα κράτη-μέλη το πρόγραμμα Εράσμους να υποστηρίζεται και από χρηματοδότηση του ΕΚΤ για ε, παιδιά και φοιτητές από πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να έχουν την ευκαιρία και εκείνοι να ε, επωφελούνται από τις διάφορες ευκαιρίες μετακίνησης των φοιτητών στην Ευρώπη. Επίσης, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο ε, Αντιμετώπισης Παγκοσμιοποίησης. Το ένα δρά έτσι κάπως προδραστικά Ε, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο φροντίζει να μην απολύονται οι εργαζόμενοι με αύξηση των προσόντων και των δεξιοτήτων του. Ενώ το Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση ασχολείται κυρίως με απολυμμένους, με μέτρα συγκεκριμένα, κομμένα και ραμμένα στα μέτρα του καθενός για να μπορέσουν γρήγορα να ξαναμπούν στην αγορά εργασίας. Στον κανονισμό έκτηση τονίζουμε και τη σημασία της εταιρική σχέσης. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν κατάλληλη και σωστή ε, συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των οργανώσεων. Και όσοι ασχολούνται ή όσους αφορά ε, η πολιτική αυτή η κοινωνική ε, προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλούμε τα κράτη-μέλη να αφιερώσουν σε κάθε πρόγραμμα τη σωστή χρηματοδότηση έτσι ώστε να εκπαιδεύουν και τους φορείς αυτούς ε, βέβαια χωρίς να τους υπαγορεύουμε τι θα κάνουν, γιατί η κατάσταση διαφέρει από χώρα σε χώρα. Ο κοινωνικός διάλογος, η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, η δυνατότητα που έχουν οι κοινωνικοί οι διάφοροι να συμμετέχουν. Απλώς ε, εφιστούμε την προσοχή στα κράτη-μέλη ότι πρέπει να συνεργάζονται με την κοινωνία των πολιτών και τους ενδιαφερομένους έτσι ώστε τα μέτρα και οι πολιτικές ε, στον τομέα που μας αφορά να πιάνουν τόπο. Έχουμε και ειδική απέτηση από τα κράτη-μέλη και μεγαλύτερο ποσοστό σε χρηματοδότησης ακόμα όταν τα κράτη-μέλη σχεδιάζουν μέτρα καινοτομίας ε, κοινωνικής και εφαρμοστικά μέτρα η κοινωνική καινοτομία δεν έχει κανένα φοβερά περιοριστικό ή σαφή ορισμό. Αυτό μπορεί να αφορά την παιδεία, την εργασία, την κοινωνική ένταξη και σχετικές δραστηριότητες. Υπάρχει χώρος για κοινωνική καινοτομία παντού στα διάφορα μέτρα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Εάν λοιπόν τα κράτη-μέλη κινηθούν προς την ανακατεύθυνση αυτή, θα έχουν αυξημένο ποσοστό συγχρηματοδότηση για προώθηση και ενίσχυση αυτών των μέτρων. Ε, ε, Επίση, εκτό από την κοινωνική καινοτομία υπάρχει και ο κοινωνικό πειραματισμό. Για να δούμε ποια είναι τα προγράμματα που υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα δεν ισχύει αυτό παντού. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σήμερα ε, έχει κάποια αποτελέσματα και κάποια συμπεράσματα που βγαίνουν από τα προγράμματα, τα οποία δεν υιοθετούν τα κράτη-μέλη, τουλάχιστον δεν τα έχουν υιοθετήσει μέχρι τώρα. Εμείς προσπαθούμε λοιπόν να ενώσουμε όλα αυτά τα νήματα, τους άξονες, ε, για να υπάρχει καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, ε, σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα για την υγεία, έχουμε ε, άμεση και έμεση εφαρμογή με 10 επιχειρησιακούς στόχους. Συνεχίζουν τις νέες προτεραιότητες που έχουν εντοπιστεί στο πρόγραμμα EASY. Συνενώνουμε τα διάφορα προγράμματα, πρώην ε, ε για να αξιοποιούμε καλύτερα και τη μικροδανειοδότηση και τη μικροχρηματοδότηση καλύτερα. Και αυτό το σκέλος του ΕΚΤ στο μέλλον θα ενταχθεί στο πρόγραμμα InvestEU με εγγυήσει ε, για τον προπολογισμό, για τις επενδύσεις σε μεγαλύτερα έργα. Θα υπάρχει και μια θηρίδα, ε, ένα σκέλος μάλλον που θα αφορά τις κοινωνικές επενδύσεις και θα εξασφαλίζει μέσω των εγγυήσεων ε, επενδύσεις στις κοινωνικές υποδομές και στις κοινωνικές δομές και στις κοινωνικές επιχειρήσεις. The health αυτός ο κλάδος της υγείας λοιπόν έχει και συγκεκριμένους στόχους επιχειρησιακούς. Είναι η συνέχιση των σημερινών ε, στόχων και προτεραιοτήτων, υποστηρικτικές δράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο που συνεισφέρουν στο να σχηματιστούν και να στηθούν στα κράτη-μέλη αποτελεσματικά, στιβαρά και ανθεκτικά συστήματα υγείας να προστατεύονται από διασυνοριακές απειλές για την υγεία και να υποστηριχθεί η νομοθεσία για την υγεία. Έχουν κοινό προγραμματισμό και παρόμοιες ομάδες στόχου. Γενικά, ε, ο κλάδος υγείας συμμετέχει στο ε, αναθεωρημένο ΕΚΤ-ΣΥΝ. Υπάρχουν κάποιε επιλέξιμες δράσεις που είναι ακριβώ οι ίδιες, αναλυτικές δραστηριότητε, εφαρμογή πολιτικής, δημιουργία ικανοτήτων, επικοινωνία και διάδοση. Και το γεωγραφικό επίση πεδίο που καλύψουν είναι αντίστοιχο με μία διαφορά. είναι επιλέξιμες όλες οι χώρες μέλη υποψήφιες και ενδεχομένε υποψήφίε, όπως τα μέλη του ΕΟΧ, οι χώρες υποπροσχώρηση, υποψήφιες χώρες και πιθανές υποψήφιες και άλλοι διεθνείς οργανισμοί, άλλες τρίτες χώρες. Ενώ για το κλάδο της υγείας έχουμε και τη χώρα της, χώρες που είναι επιλέξιμες, ακριβώς για να εξασφαλίσουμε ότι οι απειλές στην υγεία δεν συνοριακές λαμβάνονται ε, υπόψη και αντιμετωπίζονται γιατί πολλές φορές περνάνε από τη μια χώρα στην άλλη. Υπάρχει και ένα άρθρο για τις επιτροπές Υπάρχει μια επιτροπή ε, το άρθρο 163 της ε, ε, ΣΛΕ, Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία επιτροπή αυτή θα παρακολουθεί την υλοποίηση όλων αυτών των κλάδων του ΙΣΕΦ-ΣΥΝ. Η, η Επιτροπή Επιτροπολογίας για το ενισχυμένο ΕΚΤ, επιμερισμένη διαχείριση, είναι αυτό που είναι αυτή που θεσπίστηκε από το μελλοντικό κανονισμό περί κοινοδιατάξεων. Οπότε έχει νόημα να έχουμε μία και μόνο επιτροπή για όλα τα προγράμματα που πληρούν τους ίδιους κανόνες εφαρμογής ε, που προβλέπει ο κανονισμός περί κοινών Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας και είμαι έτοιμη για τη συζήτηση. Πολύ ευχαρίστω να απαντήσω και στις απορίες σας, ερωτήσεις σας. Και νομίζω ότι η σημερινή συζήτηση θα είναι μια πολύ καλή βάση για τις μελλοντικέ μας διαπραγματεύσεις. Ευχαριστούμε κυρία Σούκοβα. Πολύ καλή αυτή η εισαγωγή που μας κάνατε στο νέο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ, το ενισχυμένο. Όλοι έχουμε επίγνωση εδώ στην αίθουσα, στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα. Και μάλιστα είναι τόσο ενδιαφέρον που διεκδικούν τις αρμοδιότητες για το θέμα, για το πρόγραμμα αυτό και άλλες επιτροπές. Πάντως η απασχόληση και τα κοινωνικά θέματα είναι δική μας αρμοδιότητα και θα την διεκδικήσουμε με επιμονή. Και δεν θέλουμε κανένα διαχωρισμό μεταξύ των δύο σκελών της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων. Θέλουμε να μείνουν μαζί. Ε, πολύ χρήσιμη αυτή η γενική επισκόπηση που μας κάνατε για την πρόταση για το νέο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το διευρυμένο ή ενισχυμένο. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Λόπε Φοντανιέ, την εισηγήτριά μας για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίαση που μας έκανε και όπως είπε και η Πρόεδρος μας, ήταν πολύ σαφής, ξεκάθαρη και μας έδωσε μια γενική ε, εικόνα για τη νέα πρόταση που θα μας βοηθήσει πολύ και στην εκπόνηση των τροπολογιών στη συνέχεια. Πριν προβώ σε μια αξιολόγηση της πρότασης, θα ήθελα να σας αναφέρω κάποιο προβληματισμό μου για το Ταμείο Περικοινών Διατάξεων και πώς θα επηρεάσει το νέο ενισχυμένο ΕΚΤ, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη μείωση της ε, χρηματοδότησης, ε, την, την κατάργηση ουσιαστικά της προκαταβολής της και την πρόταση να περάσουμε από το νησιν 3 στο νησιν 2, κάτι που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα τα οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Και έρχομαι στο κυρίω θέμα. Γενικώ ε, ενστερνίζομαι τους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την καλύτερη σύνδεση του ενισχυμένου ΕΚΤ με τις ειδικές συστάσεις αναχώρα, αλλά και με τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Θα πρέπει να αποδείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, φέρνει τα κοινωνικά ζητήματα στο επίκεντρο της πολιτικής της. Αυτό είναι πολύ σημαντικό μήνυμα. Και μάλιστα ε, εστιάζεται και στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και προτείνεται συγχώνευση διαφόρων ταμείων και προγραμμάτων σε ένα ενιαίο διευρυμένο ΕΚΤ. Ε, έτσι θα πλουστεύσουμε, πιστεύω, τις διαδικασίες, όπως είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα διευκολύνουμε την υποβολή αιτήσεων για κονδύλια και θα ε, εφαρμόσουμε μεγαλύτερη ελαστικότητα ώστε τα επιχειρησιακά προγράμματα να προσαρμοστούν στις ανάγκες και να αντλούν κονδύλια από διάφορα ταμεία. Πάντως αυτή η συγχώνευση με προβληματίζει κάπως και με ανησυχεί, γιατί κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε να διατηρήσουμε τους συγκεκριμένους μας στόχους όπως την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων ή την εξάλληψη της φτώχειας. Δεν ε, μπορούμε να δεχτούμε αλλίωση των στόχων αυτών, η άμβλησή τους. Η πρωτοβουλία για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων ήταν ε, πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Γιατί α, εστιάζεται σε άλλο σημείο, γιατί ξεκινούσαμε από μία περιφερειακή επικέντρωση ε, και εσείς προτείνετε μια εθνική τώρα εστίαση. Μήπως αυτή η μεταστροφή αποβεί βάρος ε, των περιοχών που έχουν πληγεί περισσότερο από την ανεργία των νέων. Γιατί αν η χώρα στην οποία ανήκουν δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για τη χρήση των 10% των κονδυλίων, θα πληγούν αυτές οι περιφέρειες. Επίσης, ε, μην ξεχνάτε ότι χώρες με, τη, με τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας των νέων έχουν και πολύ μεγάλα ποσοστά ανεργίας του γενικού πληθυσμού, οπότε έχουν πολύ πιο δύσκολη οικονομική κατάσταση. Και διαπιστώσαμε ότι τα κράτη-μέλη έχουν προβλήματα για την ε, θέσπιση των, και εφαρμογή των εθνικών τους προγραμμάτων. Πολύ φοβάμαι ότι το ίδιο θα γίνει ε, από τη στιγμή που θα καταργήσουμε την προχρηματοδότηση και ταυτόχρονα με την πρόταση αύξηση ε, του ποστού συγχρηματοδότηση, δηλαδή του εθνικού μεριδίου στη συγχρηματοδότηση, θα ε, ενταθούν τα προβλήματα, γιατί ακριβώ οι χώρε που έχουν οικονομικά προβλήματα καλούνται να αυξήσουν τι προσπάθειέ του. Επίση, με ενδιαφέρει η καταπολέμηση τη φτώχεια και του κοινωνικού αποκλεισμού. Χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει 25% των κονδυλίων του ΕΚΤΣΙΝ να αφιερωθούν στο στόχο αυτό. Δεν αρκεί όμως αυτό το ποσοστό. Πολλό δε μάλλον που το Ευρωπαϊκό Ταμείο Βοήθειας στους Απόρους έχει συγχωνευτεί στο νέο έκτηση. Γι' αυτό θα έλεγα το 2% που προβλέπεται για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Βοήθειας σε Απόρους να προσθεθεί στο 25%, δηλαδή να έχουμε 25 συν 2%. Γιατί οι δικαιούχοι, οι άποροι δηλαδή, χρειάζονται βοήθεια για να ορθοποδήσουν στις ευρωπαϊκές χώρες και μάλιστα σε όλες τις χώρες, άσχετα από το επίπεδο φτώχειας ε, και κοινωνικού αποκλεισμού που έχει κάθε χώρα. Ένα άλλο σημείο που θα ήθελα να επισημάνω είναι η τα άτομα με αναπηρίες. Πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε ρητή μνήα στην έκθεση ε, της ε, των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Γιατί θα... δεν θα καταφέρουμε να εγγυηθούμε τη σωστή εφαρμογή των κονδυλίων με βάση τις δεσμεύσεις μας που απορρέουν από τη σχετική σύμβαση του ΟΗΕ, που ήδη έχει κυρωθεί από όλα τα κράτη-μέλη. Και τέλος, ένα θέμα που κατά τη γνώμη είναι πολύ σημαντικό, είναι η σύνδεση με το άρθρο 174 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ και χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, το στόχο της αηφόρου ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς. Αν όμως ε, επικεντρωθούμε μόνο στις οικονομικές και τις κοινωνικές πτυχές, ξεχνώντας την εδαφική διάσταση που είναι σημαντική για να αντιληφθούμε τη λειτουργία σε συγκεκριμένη περιφέρεια, δεν θα καταφέρουμε τους στόχους μας. Είπατε ότι επικεντρώνεστε κυρίως στις εξόχως απόκεντρες περιοχές ή τις ε, βόρειες περιοχές ή σε άλλες περιοχές που έχουν δημογραφικά, ε, ή, όχι, όχι όμως σε άλλες περιοχές που έχουν μόνιμα δημογραφικά ή άλλα προβλήματα. Η δική μου περιφέρεια, η Αραγών στην Ισπανία, παρόλο που θεωρείται ανεπτυγμένη, αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα αεροκατοικημένου πληθυσμού και στη φιλία. Στο μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού βρίσκεται στην πρωτεύουσα. Αν το συνδυάσουμε αυτό με τη γύρεση του πληθυσμού που είναι πολύ εντονότερη στι αγροτικές ζώνες, αντιμετωπίζουμε μια πολύ κρίσιμη κατάσταση και το μεγαλύτερο τμήμα τη Αραγών ε, απειλείται με εμφανισμό. Δεν είναι μόνο αυτή η περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Αραγώνια και άλλες περιφέρειες έχουν αντίστοιχα προβλήματα. Έχετε κατά νου κάποια προβλήματα μέτρα ε, για να προτείνεται για τις περιφέρειες αυτές, αντίστοιχα με αυτά που προτείνεται για τις ιδιαίτερα ε, βόρειες περιοχές της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρόλο που δεν έχουν παρόμοια προβλήματα, δεν έχουν τέτοια προβλήματα, αλλά έχουν εξίσου δύσκολα προβλήματα. Κυρία Γιονγκέρης, μου επιτρέπετε να δώσω πρώτο λόγο στην κυρία Τσίμερ που είναι σκιώδη συγγήτρια, πριν να το δώσω εσάς. Καλώς. Κυρία Τσίμερ που είναι και σκιώδη συγγήτρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε τον λόγο και το μικρόφωνο. Να σας ευχαριστήσω για την ε, παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ΣΥΝ. Ε, έχει πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία το θέμα της ενοποίησης των ταμείων και προγραμμάτων Επί της αρχής ε, βεβαίως είναι σωστό αυτό για να αποφύγουμε διπλές ενισχύσεις, αλληλεπικαλύψεις κτλ. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι πρέπει να προσέξουμε ε, ότι τα ταμεία αυτά έχουν τις δικές τους ε, συγκεκριμένες αποστολές που δεν πρέπει να ξεχνάμε και πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία βεβαίως μιας ισχυρότερης συνεργασίας και ενοποίησης. Ταυτόχρονα θα ήθελα να πω ότι ε, ήταν ενδιαφέρον αυτό το οποίο μόλις είπε η συγγήτρια. Θεωρώ ότι μας περιγράφεται μια κατεύθυνση εργασίας που θα μπορούσε να είναι πολύ σημαντική για εμάς στις ε, συζητήσεις των σχεδόν εισηγητών και οπωσδήποτε θα προσεγγίσουμε σε διάφορα ζητήματα. Θα ήθελα όμως να αναφερθώ σε κάτι ακόμα. Συζητάμε για την εμπλοκή ιδιωτικών φορέων και βεβαίως ε, αυτό έχει σκοπό την καλύτερη χρηματοδότηση έργων και προγραμμάτων. Έχω όμως τον φόβο ότι ειδικά στον κοινωνικό τομέα, καθώς έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους οι οποίοι δεν εντάσσονται έτσι πάρα πολύ απλά σε κριτήρια οικονομικής αποτελεσματικότητας, ε, γέρεται το ερώτημα σε ποιο βαθμό θα μπορούσε κάποιος να επηρεάσει την κατεύθυνση των προγραμμάτων, των έργων. Αυτό είναι σημαντικό, καθώς σε περιφερειακό επίπεδο οι εταίροι οι οποίοι συνεργάζονται εκεί πέρα γνωρίζουν ε, και ποια είναι τα συγκεκριμένα προβλήματα και λένε αυτό είναι σημαντικό για εμάς. Οπότε θεωρώ ακριβώς ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και θα ήθελα να μας πείτε κάπως πιο συγκεκριμένα πώς θα αποφευχθεί κάτι τέτοιο για να υπάρχει αυτή η δημοκρατική συμμετοχή των ε, εταίρων. Αυτό ήθελα να πω, οπωσδήποτε τα άλλα θα τα βρούμε μετά στη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσω τον λόγο στην κυρία Τρεμπέσιους από το ECR. Έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εκπρόσωπο της Κομισιόν για την αναλυτική της ε, παρουσίαση. Έχω αντιληφθεί βεβαίως ότι έχουμε διαφορετικά προγράμματα τα οποία προσπαθείτε να ενοποιήσετε και να απλοποιήσετε και αυτό είναι κάτι το οποίο οπωσδήποτε η ομάδα μας χαιρετίζει. Θέλουμε μια πιο αποτελεσματική Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα δεν ξέρω αν οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν με τα προγράμματα τα οποία παρουσιάζεται. Έχουμε αμφιβολίες για το ότι εάν το μεγαλύτερο περιθώριο ευελιξίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα χρησιμοποιηθεί για να ανακατευθυνθούν τα χρήματα από βόρα προς νότον για να σταθεροποιηθεί το ευρωσύστημα. Βλέπουμε ότι οι πληρωμές προς την Γερμανία θα περικοπούν στο νέο πι και ε, θα έχουμε μία συνέχεια των όσων είδαμε στην λεγόμενη διάσωση του ευρώ. Οπότε θα πληρώσει τρεις φορές η Γερμανία τον Brexit. Μεγαλύτερες πληρωμές, λιγότερες επιστροφές και βεβαίως μία μεγαλύτερη ε, βλάβη της ε, γερμανικής οικονομίας καθώ ήταν περισσότερο διαπεπλεγμένη με την Βρετανική. Και μιλάτε επίσης για τα συγκεκριμένα άτομα τα οποία είναι μειονεκτικά και μιλάτε εκεί μέσα για πρόσφυγες και μετανάστες. Εδώ πέρα έχουμε πολιτικούς στόχους που επισέρχονται, πρέπει να χωριστούν αυτά τα δύο. Και μετά μιλάτε για τις, τους επιπρόσθετους στόχους ε, που πρέπει να επιτύχουν τα κράτη, αλλά δεν το κάνουν. Τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα όμως για τα συστήματα εκπαίδευσης. Πρέπει λοιπόν να αναμένουμε από τα κράτη να αναλαμβάνουν αυτές τις ε, ευθύνες τους. Δεν είναι δυνατόν αυτά να τα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 194 να περιορίζεται σε αυτά τα οποία τις αναλογούν. Θεωρούμε λοιπόν συνολικά ότι το έκταση είναι ε, κάτι το θετικό, αλλά θα θέλαμε να υπάρχει κάποια μεγαλύτερη ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Θα δώσω τον λόγο στην ε, κυρία Γιονγκέριου από σοσιαλδημοκράτα. Σοσιαλδημοκράτες. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ και την ε, Κομισιόν. Εγώ αντικαθιστώ την ε, δική μας την εισηγήτρια. Ελπίζω την παρουσίαση αυτή να μας την δώσετε γιατί θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη και για τις συζητήσεις στην πολιτική μας ομάδα. Ο Μπράντο μου ζήτησε να κάνω κάποιες παρατηρήσεις εκ μέρους του. Το νέο αυτό Εκτασίν ε, σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παραμείνει ανταγωνιστική στην οικονομία με το να διασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο απασχόλησης, εκπαίδευση υγεία κοινωνικής ένταξη και ως σοσιαλιστές και δημοκράτες θεωρούμε ότι αυτό είναι μια προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, τα χρόνια που έρχονται και άρα θα παίξει ένα κρίσιμο ρόλο για να έχουμε έναν μηχανισμό ο οποίος θα λειτουργεί. Το ΕΚΤΣΥΝ τώρα θα είναι το βασικό μέσο εφαρμογής του πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. αλλά χρειάζονται κάποιες ε, διευκρινήσεις. Η σημαντικότερη διευκρίνηση αφορά την σχέση μεταξύ του ΕΚΤ ε, ΣΥΝ και των ε, συστάσεων αναχώρα γιατί πώς ε, μπορούμε, και αυτή είναι η ερώτησή μου, να διασφαλίσουμε ότι μέσω της διαδικασίας του εξαμήνου οι συστάσεις αυτές πραγματικά θα αφορούν τις κοινωνικές ανάγκες στα κράτη-μέλη. Πώς μπορούμε να αγγίσουμε κάτι τέτοιο. Δεύτερον, η Κομισιόν προτείνει το κατάλληλο ποσό τα κονδυλίων που θα πρέπει να δοθεί στο πλαίσιο των στόχων αλλά αυτό κατά την άποψή μας μοιάζει σαν να δίνει ένα περιθώριο διακριτικής ευχέρειας γιατί βεβαίω ε, με αυτή τη διατύπωση μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει και να δημιουργηθεί ένας ε, βαθμός αβεβαιότητας για τον προγραμματισμό των πόρων. Όχι μόνο για το πόσα λεφτά ε, σημαίνει, αλλά και το ποια μέτρα θα χρηματοδοτηθούν. Τέλος, υπάρχει μια ουσιαστική αλλαγή όσον αφορά την καταπολέμηση της ε, ανεργίας των νέων. Και βεβαίω αυτό είναι κάτι το οποίο μα είναι ιδιαίτερο αγαπητό. Όταν λοιπόν αυτή η πρωτοβουλία εξαφανιστεί για τους νέους και θα έχουμε απλά ένα 10% στις σχετικές δράσεις για την ανεργία των νέων. Πώς ακριβώς, αυτή τη διευκρίνηση ζητάω, πώς θα εγγυηθούμε ότι θα υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση για τον στόχο αυτό που όπως είπα μας είναι ιδιαίτερος αγαπητός. Πώς θα διασφαλίσουμε ότι η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων θα παραμείνει προτεραιότητα και δεν νομίζετε ότι χρειαζόμαστε να ενισχύσουμε τις αναφορές στον στόχο για την εγγύηση για την νεολαία που είναι πολύ περιορισμένες. Και να κάνω και μια δικιά μου ερώτηση εισηγήτρια για τις ε, προτάσεις αυτές. Στα τελευταία σας διαφάνεια μιλήσατε για επιτροπολογία. Τι κάνουμε. Πώς θα εγγυηθούμε δηλαδή με αυτήν την διαδικασία, την σφραγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν όλα αυτά θα πάνε στην επιτροπολογία μήπως ε, ε, έπρεπε να εγγυηθούμε ότι θα εμπλακεί και το Κοινοβούλιο. Α, και το Συμβούλιο βεβαίω, αλλά στα πόνα ήδη Για την διαχείριση των κονδυλίων, ευχαριστώ. Thank you very much. <coughs> Sorry. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω κανέναν να εκπροσωπεί την ομάδα των φιλελευθέρων. Απουσιάζει. Οπότε ακολουθεί η κυρία Λάμπερτ, εξ ονόματος των Πρασίνων, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω εξ ονόματος της Τέρι και που είναι η δική μας και ηγετρία. Θα ήθελα πάρα πολύ να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίαση. Και παρακαλώ να τη λάβω, γιατί δεν τα συγκράτησα όλα αυτά. Θα σας ήμουν ευγνώμων να μας τη δίνατε. Επίσης, ε, για την ανάπτυξη δεν έχουμε μόνο την έξυπνη ανάπτυξη, έχουμε και την πράσινη ανάπτυξη και καλό θα ήταν να φέρετε αυτό έτσι κάπως πιο στεναρά στην, ε, στη διαφάνεια και όχι εν παρόδο. Θέλω να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια γιατί υπάρχουν κάποια σημεία όπου πραγματικά συμφωνούμε. Να πω δύο λόγια για το την κοινωνική ένταξη και το κονδύλι 25% που έχετε προσημειώσει. Είναι πολύ θετικό. Είναι άραγε και επαρκές. Ε, αυτό είναι συζητήσιμο. Αν θέλετε μπορούμε να το συζητήσουμε. Ανησυχούμε επίσης για τον τρόπο με τον οποίο η βοήθεια και το Ταμείο για τους Απόρους έχει ενταχθεί τώρα ε, μέσα σε αυτό το 25%. Για ποιο λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πήρε το 2% ως μέσο για 4%. Ε, τα κράτη-μέλη είναι τόσο διαφορετικά στην αντιμετώπιση όπου το, το 2% του θεωρείται κατάλληλο και πού θα, θα, βρείτε αυτά τα χρήματα ε, και είναι ενδιαφέρον να το συζητήσουμε με αυτό με την εισηγητρία. Επίσης μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να δούμε να ευθυγραμμίζονται πολύ περισσότερο αυτές οι διαδικασίες με τις στάσεις αναχώρα, με τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ακριβώς για να αποκτήσουν και μεγαλύτερο ειδικό βάρος οι συστάσεις για τα κοινωνικά θέματα. Αυτό είναι σημαντικό για μας και με τον πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων και τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Όλα αυτά όμως κάπως θα πρέπει να είναι και πιο ορατά και να προβάλλονται, φαίνονται δηλαδή στο ΕΚΤ συν το ενισχυμένο. Θα κάνουμε τροπολογίες προς την κατεύθυνση αυτή. Και κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες θέλουμε. Να, <laughs> έχουμε διδαχθεί από τις χείριστες, όχι τις βέλτιστες πρακτικές ορισμένων κρατών μελών. Ε, συνέχεια μιλάμε για τις καλές και τις βέλτιστες, να μην ξεχνάμε και τις κακές πρακτικές και να μην υποστηρίζονται εκείνοι που παραβιάζουν το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων και των πυλών ε, των κοινωνικών δικαιωμάτων. Χαίρομαι που επαναλαμβάνετε ότι σας ενδιαφέρουν τα θέματα ισότητας, τα σχετικά θεματολόγια κατά των διακρίσεων και δεν υποστηρίζονται δράσεις που οδηγούν σε κοινωνικό διαχωρισμό, ακόμα και κοινωνικό αποκλεισμό. Αυτό το έχουμε δει πολύ έντονο στο σημερινό πρόγραμμα για άτομα με αναπηρίες. Επίσης, τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε για να υπάρχει καλύτερη πρόσβαση και πιο εύκολη για μικρότερους φορείς και οργανώσεις. Θα κάνουμε και εκεί τροπολογίες για να ενισχυθεί η εταιρική σχέση και η σχετική αρχή. Βασικά το θέμα είναι τι ρόλο διαδραματίζει η κοινωνία των πολιτών σε αυτά τα ζητήματα. Και έχω και μια ερώτηση για το σημερινό άρθρο 40 εδάφιο 2. Αυτά είναι τη Στέρι Ράιντ και όλα που σας λέω. Για ποιο λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει συμπεριλάβει κοινωνικές οργανώσεις ε, ε, ως παρατηρητές ε, στην, στις επιτροπές Αυτό το καθεστώς το έχουν ήδη. Γιατί δεν το αναφέρετε ρητά στο νέο κανονισμό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν και άλλοι τομείς και πολλοί που θα καταθέσουμε τροπολογίες, αλλά προς το παρόν αυτά ήταν κάποια ερωτήματα και κάποια θέματα που ήθελα να θέσει κύριε Ρέντ και η Πράσινη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καλδές, Καλβές Σαμπόν εκπροσωπείται του σκιώδη ηγετή του των Φιλελευθέρων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Ελίμοβιτς είναι ο αρμόδιος και ο αλλά ε, ασθενή και απουσιάζει. Η ιδέα ε, συγχώνευση των προγραμμάτων σε ένα είναι γενικά καλό για μας ε, τους φιλελευθέρους. Θα πρέπει να έχουμε αποτελεσματικότητα, απλούστευση, συνέργεια και τα ταμεία να εκτελούνται σωστά, με ευελιξία στις εθνικές συνθήκες, στις δυνατότητες κάθε χώρα και στις ανάγκες κάθε χώρας η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και δυναμικό είναι πάρα πολύ σημαντική για μας. Άλλο σημαντικό για μας είναι ε, η μη διάκριση στις ευκαιρίες σε πιο έξυπνη Ευρώπη, πιο πράσινη Ευρώπη και με λιγότερο διοξίδι του άνθρακα. Ανησυχώ για την πρωτοβουλία ε, για την ε, ασχόληση των νέων. Φαίνεται ως ξεχωριστό ταμείο δεν πήγε καλά, οπότε θα πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα για να γίνει μια πραγματική αλλαγή. E ε, αυτό που θέλουμε είναι να δούμε το έκτηση να ευθυγραμμίζεται με το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Και αυτή τη γραμμή θα ζητήσουμε από πλευράς φιλελευθέρων να ακολουθηθεί άλλη τεράστια πρόκληση μπροστά μας είναι το Brexit. Άρα χρειαζόμαστε περισσότερες συνέργειες με δημιουργίες δυνατοτήτων, έρευνα, κινητικότητα εργαζομένων, ασφάλεια και μετανάστευση και να μην ψάχνουμε τώρα νέες προτεραιότητες. Σε ό,τι αφορά το Ταμείο για την ενίσχυση των απόρων, θα πρέπει αυτό να παραμείνει συμπληρωματικό προς τη, τα διάφορα συστήματα που υπάρχουν στα κρατημέλη, χωρίς να τα υποκαθιστά ή να τα αντικαθιστά χρειάζονται συνοδευτικά μέτρα για την ηλική υποστήριξη. Ας πούμε, όλοι κάνουμε ε, τέτοια κινήσεις. Αν στέλνουμε, στέλνουμε όμως δέματα με τρόφιμα, αντιμετωπίζουμε μια σημερινή ανάγκη, αλλά δεν λύνουμε το πρόβλημα. Αυτό το θέμα του κοινωνικού αποκλεισμού και της κοινωνικής ένταξης είναι πολύ σημαντικό και προσωπικά ε, είμαι υπέρ της ένταξης των μεταναστών των Ρωμά και πολιτών των κρατών. Παρ' ε, όλα αυτά θα πρέπει να έχουμε υπόψη και τις εθνικές αρμοδιότητες ό,τι αφορά το σκέλος της υγείας. Θα πρέπει να σεβόμαστε τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες των κρατών μελών για τις πολιτικές υγείας και το πώς θα οργανώνουν και πώς θα παρέχουν ε, την υγεία και τις φροντίδες υγείας. Εμείς να συνοδεύουμε και να συμπληρώνουμε ε, τις εθνικές πολιτικές πάντα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού Αλλά η χρηματοδότηση και η οργάνωση των συστημάτων υγείας θα πρέπει να παραμείνουν αρμοδιότητα των κρατών μελών. Και τέλος, περιμένω εδώ το σχέδιο έκθεσης και να το συζητήσουμε. Και οπωσδήποτε θα κάνω και τροπολογίε. προς τη γραμμή αυτή των φιλελευθέρων. Με επικοδομητικό πνεύμα όμως. Αξίζει να αναλύσουμε αυτή την προσπάθεια που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είμαι βέβαιος ότι η συγκήτρια ε, θα κάνει προσπάθειες για να τη βελτιώσει και μόνο. Σας ευχαριστώ. Δεν βλέπω κανένα από την ομάδα EFTD. Κυρία Λάουρα, άτζεα κανονικά. Αλλά δεν βλέπω και κανέναν από την ομάδα ENF. Μάλιστα. Θέλετε κυρία Φοντάνιε να δευτερολογήσετε. Δεν χρειάζεται, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Προτιμώ να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλώ ήρθατε να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω ε, τα μέλη που έλαβαν το λόγο. Σίγουρα η ενεργεία των νέων είναι η πρωταρχή προτεραιότητα όλων μας και θα φροντίσω να παραμείνει και στην προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, θέλουμε να απλουστεύσουμε την εφαρμογή, γιατί έχουμε επικριθεί μέχρι πρόσφατα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι ο ρυθμός εφαρμογής δεν είναι αρκετά ταχύς. Θα πρέπει να προσφέρουμε πιο άμεση βοήθεια σε όσοι είναι εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης και να ε, βελτιώσουμε την ένταξη των ε, νέων στην αγορά εργασίας. Και σίγουρα δεν ακυρώνουμε την πρωτοβουλία για την ενέργεια των νέων, αλλά απλώ ε, ε την εντάσσουμε σε αυτό το ε, νέο ενισχυμένο πρόγραμμα, το ECT-SYN, και επίσης έχουμε προσθέσει κάποια κριτήρια στα πλαίσια της παρακολούθησης ε, των συστάσεων για την εγγύηση των για τους νέους σε ό,τι αφορά τη βιότητα των προσφορών που έχουν εντοπιστεί και παρουσιαστεί υποβληθεί στους νέους άσχετα από το αν χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς προπολογισμού, ή το κονδύλιο για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Και συνεχίζουμε την συνεργασία με τα κράτη-μέλη για να βελτιωθούν οι πολιτικές τους για τους νέους και να μπορέσουν τα κράτη-μέλη πραγματικά να αγγίξουν τους νέους που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης, απασχόληση και να τους βοηθήσουν να επανέλθουν είτε σε εκπαίδευση είτε σε απασχόληση. Ε, και το ότι δεν είναι η πρωτοβουλία για τους νέους ε, ε, ξεχωριστό κονδύλιο και συγχωνεύεται με το ΕΚΤΣΙΝ δεν θα υπονομεύσει ούτε θα υποτιμήσει αυτή την πρωτοβουλία. Επίσης είπαμε ότι υπάρχει δυνατότητα και για τα κράτη-μέλη που έχουν τα 10 που έχουν το 10% και λέμε τουλάχιστον το 10% το κονδύλιο του ΕΚΤ στο μέλλον χρησιμοποιηθεί για την ανεργία των νέων. Δηλαδή δεν θα είναι λιγότερο από 4,4 δις ευρώ. Οπότε έχουμε παρόμοιο κονδύλιο με αυτό που προβλέπεται και στα υποχρεωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων. Παρόλο που τα μισά κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή, ε, γιατί στους περιφερειακούς δίκτες είχαμε 20 κράτη-μέλη όταν ξεκινήσαμε το πρόγραμμα, τώρα έχουν μείνει 11. Και στο μέλλον, στο μέτρο που βελτιώνονται οι καταστάσεις, θα έχουμε 10 κράτη-μέλη. και περίπου το ίδιο κονδύλιο. Οπότε θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να φτάσουν στους πραγματικούς δικαιούχους αυτά τα κονδύλια και σε καμία περίπτωση δεν παρεμποδίζουμε ή δεν περιορίζουμε τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν κονδύλια του ΕΚΤ για να στηρίξουν τους νέους. Η αναγνώριση ε, ένα ταμείο, μία προσπάθεια δεν σχετίζεται με τον τίτλο, το όνομα του ταμείου, αλλά το στόχο, γιατί έχουμε, θέλουμε να έχουμε λιγότερο νέους ε, που να ανέργους ή που θα εγκαταλείπουν το σχολείο ή που δεν θα έχουν δεξιότητες και δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Στόχος είναι να έχουν όλοι ισότιμη πρόσβαση στην ε, απασχόληση, ανάλογα με τις σπουδέ τους και τις δεξιότητές τους. Αυτό άσχετα με τα επίπεδα ενεργείας, αν είναι ε, χαμηλότερα ή υψηλότερα από τον κοινοτικό μεσόωρο. Επίσης, πώς θα συνδυάσουμε το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, με ρωτήσατε, τον κύκλο και τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού εξάμεινου με το δικό μας προγραμματισμό και πώς ε, οι προκλήσεις που εντοπίζονται στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο αλλά και στις ε, εκθέσεις αναχώρα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με πολύ διεξοδική ανάλυση για την προετοιμασία των ειδικών συστάσεων χώρα, πώς θα ληφθούν υπόψη και θα αντικατοπτρίζουν τις προκλήσεις ε, που καλείται το ΕΚΤ να αναλάβει. Θα ετοιμάσουμε το μηχανισμό για τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του 2019 με πολύ ε, πιο διεξοδική ανάλυση που θα δίνουμε στις εκθέσεις αναχώρα και με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ποια είναι τα κυριότερα επενδυτικά χάσματα που εντοπίζουμε στα κρατη τα επενδυτικά κενά και προτείνουμε αυτά να καλυφθούν με τη βοήθεια και του κοινοτικού προϋπολογισμού. Επίσης, στις ε, ειδικές συστάσεις αναχώρα κάνουμε μνήα των ε, ε, προκλήσεων που αφορούν τα επενδυτικά κενά και αυτά τα συνδέουμε με τους σκοπούς των επιμέρους ταμείων. Και αυτό θα είναι το σημείο αφετηρίας μας για τις διαπραγματεύσεις με τις χώρες μέλη. Θα συζητήσουμε με τα κράτη-μέλη με βάση την ε, ανάλυση που κάναμε, την ενδελεχή. Και θα πούμε από τα κράτη, στα κράτη-μέλη πού περιμένουμε να αφιερώσουν τα κονδύλια και θα μας πούν και τα κράτη-μέλη ποια θεωρούν σημαντικότερες προτεραιότητές τους. Η διαδικασία των διαπραγματεύσεων των εταιρικών σχέσεων και των προγραμμάτων είναι χρονοβόρα Μερικές φορές κρατάει και μία διετία και παραπάνω ίσως. Γι' αυτό θέλουμε οι κοινοτικοί στόχοι να στηρίζονται και να χρηματοδοτούνται με κοινοτικό προπολογισμό. Όταν είναι καλύτερο αυτό το επίπεδο. Αυτό δεν σημαίνει ότι συρρυκνώνεται η επικουρικότητα ή υπονομεύεται η επικουρικότητα ούτε στις πολιτικές, ούτε στην παιδεία, ούτε στις κοινωνικές πολιτικές, ούτε στην υγεία. Έχουμε επίγνωση απόλυτη της επικουρικότητας στους τομείς αυτούς και επιτρέπουμε στα κράτη-μέλη να επενδύσουν με τα κονδύλια αυτά εκεί που πιστεύουν ότι είναι μεγαλύτερες ε, ανάγκες και που βλέπουν τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία από τη χρήση των κονδύλιων. Επίσης, βοηθούμε τα κράτη-μέλη να μην υποκαταστήσουν με τα κοινοτικά κονδύλια τον εθνικό τους προπολογισμό και το θέμα του Ταμείου των Απόρων και εκεί δεν θέλουμε να υποκαταστήσουμε τα, τις εθνικές για τους απόρους. Και γνωρίζουμε ότι 118 εκατομμύρια συμπολιτών μας βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού πριν από δύο χρόνια και δεν θα μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε ή να εξαλείψουμε τη φτώχεια με 2-3 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν πρόκειται, δεν είναι εφικτό κάτι τέτοιο, είναι τελείως τοπικό. Πάντως, στην τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού, το Ταμείο για τους Απόρους βοήθησε την αλλαγή των εθνικών πολιτικών και την αλλαγή νοοτροπία στα κρατημέλη. Ακόμη και με περιορισμένο κονδύλιο, είχαμε μια σημαντική μεταστροφή στην προσέγγιση του προβλήματος και στο πώς ε, χρησιμοποιούνται οι πολιτικές ή εφαρμόζονται οι πολιτικές απέναντι στους απόρους και τους ε, απειλούμενους από κίνδυνο αποκλεισμού. Και φυσικά με την ηλική υποστήριξη έχουμε και τη συνεργασία με ΜΚΟ που έχουν αποκτήσει πολύ πείρα και αυτοπεποίθηση από τη συνεργασία με, τις, με τους χορηγούς και χρησιμοποιούμε αυτές τις ε, ΜΚΟ, του τους εταίρους μας για να δρομολογήσουμε τις επιπλέον, τις συμπληρωματικές δωρές. Επίσης, τα κράτη-μέλη βοηθούμε και φτωχές οικογένειες ε, και βοηθούμε κυρίως τα τέκνα αυτών των οικογενειών χωρίς να τα στιγματίζουμε. Οπότε θα έχουμε μέτρα για να βοηθήσουμε τα παιδιά αυτών των φτωχών οικογενειών ότι δεν μπορούν να καλύψουν το ημερήσιο συσίτιο των παιδιών. Αυτό το καλύπτει ε, τα σχολικά συσίτια, το Ταμείο για τους Απόρους. Έτσι θα νιώσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ε, και θα νιώσουν ίση με τους συμμαθητές τους αυτά τα φτωχά παιδιά. Επίσης δεν παρέχουμε μόνο ηλική στήριξη, αλλά ζητούμε ε, και συνοδευτικά μέτρα του Ταμείου Απόρων να δοθούν σε αυτούς που λαμβάνουν την ηλική υποστήριξη, γιατί θεωρούμε ότι η βραχυπρόθεσμη υποστήριξη, που είναι υποστήριξη επιβίωση ουσιαστικά, δεν θα λύσει το πρόβλημα χωρίς συνοδευτικά μέτρα, χωρίς ε, παροχή συμβουλών, χωρίς κάποιο προσανατολισμό ε, σε αυτούς τους απόρους για το πώς μπορούν να βελτιώσουν την κατάστασή τους και την καθημερινότητά τους. Και αυτά τα συνοδευτικά μέτρα στο μέλλον θα καλύπτονται από το Act Sin στα πλαίσια της προσπάθειας ε, μείωσης του κοινωνικού αποκλεισμού. Σε ό,τι αφορά την κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση της φτώχειας, η, η πρόταση είναι για 25%. Τουλάχιστον, σήμερα έχουμε τουλάχιστον 20% των κονδύλιων των κρατών μελών για την κοινωνική ένταξη σε εθνικό επίπεδο. Έγιναν κάποιες αυξήσει στα κρατη ξεπεράστηκε σε μερικά το 20% και έχουμε περίπου 4 δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή για μέτρα που συνδέονται με το Ταμείο Απόρων. Αλλά σε αυτά τα μέτρα περι, περιλαμβάνουμε και κάποια ε, επιχειρησιακά προγράμματα που είναι αμυγός προγράμματα κοινωνικού αποκλεισμού, όχι μόνο ηλική βοήθειας. Γι' αυτό και έχουμε το 2% τουλάχιστον που προστίθεται για μέτρα που θα στηρίζουν τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Απόρων. Επίσης, ε, έχουμε επίγνωση των συζητήσεων που γίνονται για την οδηγία για την προσβασιμότητα και τις ε, διεθνείς συμβάσεις για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκε των ατόμων με αναπηρία και να εξασφαλιστεί προσβασιμότητα για όλου. Στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων, στο άρθρο 67.2, που προσδιορίζονται τα κριτήρια επιλογή, θεσπίζεται η υποχρέωση των κρατών μελών να μεριμνήσουν ώστε τα κριτήρια επιλογή λαμβάνουν υπόψη οποιαδήποτε δράση που εξασφαλίζει προσβασιμότητα, κατά πολεμά τη διακρίση και συνάδει με το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ήδη στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν περιμένουμε την έκβαση των συζητήσεων. Ε, δεν περιμένουμε την, την ανάπτυξη προγραμμάτων και κριτηρίων επιλογή από τι αρχέ διαχείριση. Αυτό είναι προαπαιτούμενο, είναι απαραίτητη προπόθεση που την κατοχυρώνει ο ίδιο ο κανονισμό περί κοινών διατάξεων. Ε, και στις αιτιολογικές σκέψεις ε, αναφέρονται οι διεθνείς συμβάσεις και το ενωσιακό δίκαιο για τον τομέα αυτό. Για την ε, ολοκληρωμένη βιώσιμη ανάπτυξη και τις εδαφικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών γνωρίζουμε πως υπάρχει διαφορετική εικόνα ακόμα και μεταξύ των περιφερειών επίπεδου ΝΑΤΣ 2 γιατί η τωρινή απόφαση είναι ότι οι περιφέρειες αυτές είναι η βάση μας για τον προγραμματισμό τέτοιων αναγκών και για τις συγκρίσεις μεταξύ περιφερειών. Και Βεβαίω, οι περιφέρειε όταν ετοιμάζουν τα σχέδια αυτά οικονομική και εδαφική ανάπτυξη θα συζητήσουμε με την Κομισιόν ακριβώ την ισόρροπη τέτοια ανάπτυξη που καλύπτει όχι μόνο τι περιφέρειε ε, σε σχέση με την προσβασιμότητά του ε, και την κάλυψη των άγκων των ανθρώπων, αλλά και την ισόρροπη ανάπτυξη τη κοινωνία ε, και του πληθυσμού. Βλέπουμε περιοχέ να ερημώνουν από ανθρώπου και δεν μπαίνουμε βέβαια στο επίπεδο των περιφερειών ε, ΝΑΤΣ 2. Ε, Έχουμε λοιπόν Έχουμε επίσης ε, τους εταίρους που συνεργάζονται στις επιτροπές ε, παρακολούθησης. Λοιπόν, οι επιτροπές αυτές περιέχουν και περιλαμβάνουν ε, τους συνεταίρους, τις οργανώσεις, την κοινωνία των πολιτών που προσωπούν τα άτομα εκείνα τα οποία επηρεάζονται περισσότερο από τα επιχειρησιακά προγράμματα. Και βέβαια ακριβώ το θέμα είναι και η ιδιοκτησία, όπω λέμε, του προγράμματο, αλλά και η άσκηση δημοκρατικού ελέγχου των δαπανών. Η Επιτροπή αυτή λοιπόν δεν αποκλεί κανέναν. Είμαστε πάντα ανοιχτοί ε, και είμαστε έτοιμοι να περιλάβουμε μέλη και με πρωτοβουλία των μέλων, όχι μόνο, μόνο με πρωτοβουλία της ε, Κομισιόν. Όταν υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να συζητηθεί, όταν πρέπει να γίνουν ανταλλαγές ε, εμπειριών. Οπότε πηγαίνουμε πέρα από το περιεχόμενο ή την ε, παρουσίαση κάποιων, και την εκπροσώπηση κάποιων μελών στην περιοχή. Τώρα δεν έχουμε συγκεκριμένα ποσά για πρόσφυγες ή για υπηκόους τρίτων χωρών. Θεωρούμε ότι η ένταξη ανθρώπων που έχουν ε, νόμιμο δικαίωμα να μείνουν σε μια χώρα δεν σημαίνει ότι πρέπει να τους στιγματίζει, να τους καθορίζει ως ε, ομάδα στόχο, να τους κατονομάζει ως ομάδα στόχο. Θεωρούμε ότι η ένταξη γίνεται καλύτερα με τους ντόπιου, αν παρέχουμε και βέβαια πρέπει να παρέχουμε επιπλέον στήριξη για επικούς τρίτων χωρών όταν έχουν ε, δικαίωμα να μείνουν ε, τουλάχιστον για τα γλωσσικά, για να αντιληφθούν πώς λειτουργούν οι χώρες κτλ αλλά αυτό δεν είναι ε, αλληλεπικάλυψη με το Ταμείο Σύλλου και Μετανάστευσης για τα κέντρα υποδοχής ή την πρώτη υποδοχή. Θέλουμε όλοι οι άνθρωποι που έχουν ε, δικαίωμα νόμιμης παραμονής να έχουν ε, ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση ε, δεν ε, θα χωρίσουμε άρα την χρηματοδότηση που πηγαίνει σε διάφορες σε κοινωνικές ομάδες. Νομίζω ότι εξήγησα λίγο το πώς ε, θα αναπτυχθούν οι στόχοι του Ευρωπαϊκού Ταμείου ΣΥΝ στο μέλλον. Βεβαίω τα κράτη-μέλη έχουν πάντα τον ε, λόγο για να πούν ε, ποιες είναι οι κατευθύνσεις, πού πρέπει να γίνουν οι επενδύσεις, ποια είναι τα κενά και βεβαίως ε, πρέπει και τα κράτη-μέλη να καθορίσουν ποιο είναι το κατάλληλο ποσό για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, που είναι βεβαίως διαφορετικό για κάθε χώρα. Έχουμε κράτη-μέλη με πολύ ε, λεπτομερείς ε, στόχους ε, και με, ή με ένα μόνο πρόγραμμα, αλλά έχουν τέσσερα προγράμματα. Οπότε δεν σημαίνει ότι όλες οι ανάγκες καλύπτονται από αυτό το ταμείο. Έχουμε και προγράμματα τα οποία δεν σχετίζονται με επενδύσεις. Έχουμε το μέσο των μεταρρυθμίσεων, όπου οι επενδύσεις ή οι μεταρρυθμίσεις μπορούν να στηριχθούν με ένα νέο μέσο για να επιτρέψουν κάποιες δαπάνες οι οποίες δεν είναι μετρήσιμες ή ε, μας επιτρέπουν να πούμε ότι χρηματοδοτούμε αυτήν την μεταρρύθμιση. Και έχουμε βεβαίως ε, και το μέσο εργαλείο, το εργαλείο στήριξη ε, των μεταρρυθμίσεων που πηγαίνει παραπέρα. Στην Επιτροπή Επιτροπολογίας λοιπόν ε, δεν έχουμε πολλές ε, πράξεις κατά εξουσιοδότηση, γι' αυτό θέλουμε να έχουμε μία Επιτροπή Επιτροπολογίας, είναι για την κοινή διαχείριση που αφορά ακριβώ ε, την κοινή διαχείριση μόνο. Μόνο αυτήν την δέσμη μέτρων. Δεν ε, αφορά τις άλλες δέσμες. Προτείνουμε η Επιτροπή αυτή να εργαστεί με ομάδες εργασίας ε, με το, τη δέσμη της υγείας και την δέσμη easy όπως λέγεται. Εκεί πέρα υπάρχει και μια ομάδα κατεύθυνσης που έχει ορίσει η Γενική Διεύθυνση Υγείας ως τον βασικό εταίρο της για να συζητά τις προτεραιότητες και τις δραστηριότητες που ορίζονται στην σχετική δέσμη. Και το ίδιο θα κάνουμε κι εμείς για την δέσμη την easy. Δεν ε, θέλουμε δηλαδή κάποιες πράξεις κατεξιοδότηση. αναφέρθηκα στην ελεύθερη πρόσβαση για μικρές οργανώσεις και οργανισμούς και αυτό ακριβώς είναι μέρος της γενικότερης προσπάθειας να υπάρξει μια απλοποίηση στην εφαρμογή των ταμείων, να έχουμε απλοποιημένες επιλογές κόστους που είναι υποχρεωτικές εντός ενός συγκεκριμένου ποσού επένδυσης. Προσπαθούμε λοιπόν να μειώσουμε το διοικητικό βάρος ε, για την εφαρμογή των έργων και για την επιστροφή των χρημάτων μέσω κάποιων απλοποιημένων επιλογών και νομίζω ότι υπάρχουν πολλές επιλογές ήδη και στον κανονισμό των κοινωνικών ε, διατάξεων που επιτρέπουν σε μικρές οργανώσεις να ωφεληθούν με λιγότερο διοικητικό βάρος, ε, βεβαίως πάντα αποδεικνύοντας σε τι ε, διέθεσαν τα χρήματα. Για τις ε, αρμοδιότητε και εξουσίες των κρατών μελών σε καμία περίπτωση θέλουμε εμείς να τις φετεριστούμε. Να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη θέλουμε, γιατί τα κράτη-μέλη αναγνωρίζουν ότι η εφαρμογή των ε, αρχών του πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων είναι δικό τους δικαίωμα και δική τους ευθύνη. Και έχουμε τώρα ειδικέ ε, διατάξεις για τον πυλώνα, γνωρίζουμε την ευθύνη τους, αλλά πρέπει να τους δώσουμε και τα χρήματα από το ΕΚΤΣΙΝ για να ανταποκριθούν σε αυτό και η Ευρώπη να γίνει πιο κοινωνική, ε, να έχει στόχο την κοινωνική ένταξη όλων των πολιτών. Δεν θέλουμε να πάρουμε κανένα την ευθύνη και τις αρμοδιότητες ε, δίνοντας βοήθεια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για όλες αυτές τις εξαιρετικές απαντήσεις και τα γεγονότα και τα στοιχεία που μας δώσατε. Προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών είναι 25 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Και προηγουμένως θα συζητήσουμε το σχέδιο έκθεση στην Επιτροπή μας 29 ε, και 30 Αυγούστου και ελπίζω να ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας τέλη Νοεμβρίου. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Μας δώσατε πάρα πολλές απαντήσεις και τροφή για σκέψη, αξιολογήσεις, πολύ σημαντικά όλα αυτά για τη δική μας δουλειά εδώ στην Επιτροπή μας. Και οι διαφάνειες που μας δείξατε τώρα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής μας και ε, μπορείτε να τις βρείτε και αμέσως μετά τη συνεδρίαση. Προσεχή συνεδρίαση 29 Αυγούστου 2018. Μην νομίζετε ότι είναι και τόσο μακριά. Προσβλέπω σε αυτή τη συνεδρίαση, αλλά προηγουμένω προσβλέπω στι διακοπέ ε, στην πατρίδα μα στον ήλιο, να ξεκουραστούμε. Ευχαριστώ και του διερμηνείς. Οι διερμηνείς ευχαριστούν την Πρόεδρο. Σας ευχαριστώ που βρίσκεστε εδώ και μας ε, υπηρετείτε στην υπηρεσία μας για να ε, κάνουμε τις συνεδριάσεις. Ε, θέλω να ευχηθώ σε όλους σας φανταστικές διακοπές καλοκαίρι. Σας ευχαριστώ.